σχετικό αίτημα στις, εκλογικές, στις αρχές διενέργειας εκλογών της χώρας, οι οποίες δεν μας έχουν δώσει και απάντηση επί του παρόντος. Θα ήθελα να πω στους... Να ενημερώσω να πως έχω λάβει 7 σχέδια ψηφίσματος. Τελειώνει εδώ πέρα η συζήτηση, η ψηφοφορία θα γίνει στο τέλος μετά τις ε, συζητήσεις. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η συζήτηση για το Αζερμπαϊτζάν. των ε, συντακτών. Θα ακούσουμε πρώτα απ' όλα τον κύριο Ρωμεβαϊρουέδα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, εκπροσωπώ την συνάδελφο την κυρία Ουλρίκε Λούνατσεκ. Πρέπει να πω πως δεν μου αρέσει πολύ ο διαγωνισμό τη Eurovision, αλλά το ότι γίνεται σε μια χώρα με τόσο δραματική κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων με απασχόλησε. Η καταπίεση τη ε, ελευθερία έκφραση ε, του δικαιώματος του συνέρχεστε είναι ασύμβατο με τι δεσμεύσει που έχει αναλάβει το Αφγανιστάν για τη δημοκρατία, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τι θεμελιώδει ελευθερίε. Οι αζερικέ αρχέ θα πρέπει να επιτρέψουν την ειρηνική διαμαρτυρία και να απαγορέψουν την παρέμβαση των αστυνομικών στο έργο των δημοσιογράφων που καλύπτουν διαδηλώσει. Αυτό είναι ε, επίση ε, σημαντικό όπως και η άμεση ε, απελευθέρωση ε, όσων κατηγορούνται για πολιτικά ε, εγκλήματα. Δικηγόρους, δημοσιογράφους, ε, ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να εκφράσω επίσης την συμπαράστασή μου στην οργάνωση Sing for Democracy που ελπίζουν πως η δική τους δράση θα συνεισφέρει στις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και στα ανθρώπινα δικαιώματα στο Αζερβαϊτζάν. επίση ανησυχώ για τις εξώσεις και κατεδαφίσεις κτηρίων σε σχέση με τα έργα που γίνονται στον Πακού για τον διαγωνισμό της Eurovision. Ζητώ από τις αζερικές αρχές να εγγυηθούν πως η οικοδόμηση νέων κτηρίων συγγραμμίζεται με τη σχετική νομοθεσία και πως η επανεγκατάσταση των ανθρώπων θα γίνει με τρόπο διαφανή και με δίκαιη αποζημίωση. Τέλος, να πω πως εκτιμώ το ότι επιτέλους το ΕΛΚ υποστήριξε το κοινό ψήφισμα καθώς κάποια στιγμή αυτό ήταν αβεβαίο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο επόμενος ομιλητής επίσης ε, ε, συντάκτης είναι η κυρία Μαρίδια Σχάκε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Καθώς κάνουν πρόβεση οι τραγουδιστές της Eurovision, ε, θυμώνεται η φωνή του ασερικού λαού. Ενώ θα βλέπουμε όλοι το σοου, δεν τυφλώνει το κόσμο από τις προβολήσεις και την προπαγάνδα. Ανησυχούμε πάρα πολύ για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και βεβαίως οι δηλώσει κυβέρνηση δεν καλύπτουν τις πράξεις της. Σήμερα, δύο αντιπρόεδροι του κόμματος Μουσαβάτ, μέλους της, ε, διεθνού, Διεθνούς, συνελήφθησαν στους δρόμους του Μπακού. Ένα από τους έξι αντιπρόεδρους μόνο κυκλοφορεί ελεύθερος. Οι άνθρωποι είναι σε κατοίκον περιορισμό, τους απειλούν οι αρχές και η Άννα Γκαράλη έχει εξαφανιστεί εδώ και δύο μέρες. Ο Αρίφα Τζίλη και ο Τρούα Βασλή και άλλοι ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων κρατούνται εδώ και ένα χρόνο. Οι άνθρωποι αυτοί θεωρούνται πολιτικοί κρατούμενοι από την Διεθνή Αμνηστία και τους λέω δεν θα σας ξεχάσουμε. Στις αζερικές αρχές θα πω εκπληρώστε τις υποχρεώσεις σας στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ και της Συμφωνίας Σύνδεσης. Θέλετε να είστε μέρος της πολιτικής γειτονίας ή όχι. Το Αζερβαϊτζάν δεν θα είναι αξιόπιστο εάν δεν τηρήσει τα συμφωνηθέντα. Τελεία. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ντεκάιζερ επίσης συντάκτης. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν από δέκα μέρες περίπου κοίταζα, έβλεπα τις ειδήσεις στο Euronews και είδα μια καταπληκτική εκπομπή για το Αζερμαϊτζάν για τη Eurovision. Τίποτα δεν είπαν για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έδειχναν ε, το Crystal Palace. Εγώ νόμιζα ότι ήταν διαφήμιση οχι λοιπόν ήταν εκπομπή ε, του Euronews. Γι' αυτό το σημερινό ψήφισμα έχει ιδιαίτερη σημασία. Εγώ δεν θέλω να μποϊκοτάρουμε την Eurovision, ούτω ή άλλω θα ήταν και δύσκολο και να το θέλαμε, αλλά πάντως... Ε, ε, γιατί δεν λέμε τα ίδια όπως για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Κίνα. Είναι μοναδική ευκαιρία. 600 εκατομμύρια τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν το Σάββατο. Είναι μοναδική ευκαιρία για να δείξουμε ότι πέρα από το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο και τα λεφτά, στο Αζερμπαϊτζάν υπάρχει και ένα άλλο πρόσωπο που είναι ιδιαίτερα προβληματικό, δηλαδή η διάσταση της ε, παραβίωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι χιλιάδες ιδιοκτήτες διαμερισμάτων σπιτιών ε, που ε, έπεσαν θύματα έξωσης για να κατασκευαστεί το Crystal Palace για τη διοργάνωση της Eurovision είναι κάτι απαράδεκτο, παρά είναι και γι' αυτό θεωρώ ότι ε, είναι πάρα πολύ καλό που συμπαρατάχθηκαν μαζί μας συνάδελφοι από το ΕΛΚ. Είναι απαραίτητο το ψήφισμα. Σας ευχαριστούμε κυρία Ντεκάιζερ και ε, θα... Ο κύριος Έγκελ θέλει να σας θέσει μια ερώτηση. Δέχεστε. ευχαριστώ απαντάει η κυρία Ντεκάιζερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα ουσιαστικά πρώτα απ' όλα να συμφωνήσω με την ανάλυση που μόλις κάνατε και θέλω να σας ρωτήσω, εφόσον είστε οι πρώτοι που τοποθετήθηκε κατά αυτόν τον τρόπο, το εξής. Δεν πιστεύετε επίσης ότι στην ουσία όταν πρόσφατα υπεψηφίσαμε την αξιολόγηση της ε, Συμφωνίας Σύνδεσης με το Αζερβαϊτζάν, τοποθετηθήκαμε σε ένα πλαίσιο που αγνοούσε και δεν συμπεριλάμβανε τίποτα από αυτά που συζητάμε σήμερα. Δεν θα ήταν πιο χρήσιμο εξ αρχή να επιμείνουμε στο ότι δεν είναι ακόμη ένα δημοκρατικό κράτος ε, το Αζερβαϊτζάν. Ε, και νομίζω ότι έχει αλλάξει η στάση μας σε σχέση με την προηγούμενη φορά που είχαμε σχέση με, την, με το Αζερβαϊτζάν. Απάντηση. Ε, κοιτάξτε, δεν, στη πολιτική μα ομάδα συζητήθηκε το θέμα και δεν θα επανεφεύρουμε τώρα τον τροχό αυτό. Θέλω να σας πω είναι ότι ε, αυτό που αντιπροσωπεύει το Αζερβαϊτζάν με ψαγωγούς φυσικού αερίου και τα λοιπά, να μην πολύ λόγο γιατί γνωρίζετε την κατάσταση εξίσου καλά. Αν είχαμε σχέσεις μόνο με πραγματικά δημοκρατικά κράτη, δεν θα είχαμε και πολλού εταίρου. Εγώ θέλω να σας πω ότι αυτό το θέμα είναι μόνη ιδέα για μας και θα παραμείνει και κάποια στιγμή η φιλοδοξία εδώ στην Ευρώπη είναι να συνδέσουμε επιτέλους τα εμπορικά ζητήματα μαζί με τα ζητήματα δημοκρατίας. Και κάθε φορά βρίσκουμε λεπτέ ισορροπίε. Σα ευχαριστούμε και από του συντάκτε, η κυρία Μακόβη, τελευταία ομιλήτρια. Ευχαριστώ. Η περίπτωση των τριών ακτιβιστών που γνωρίζουμε αποτελούν ε, παραδείγματα καταστολή στο Αζερβαϊτζάν. Θα ήθελα να καταδικαστούν οι πέτοι και επίσης να δούμε κατά πόσο υπάρχουν παράνομες κρατήσεις κατά των ε, διαδηλωτών και αυτή την εβδομάδα. Θα πρέπει να, να απελευθερωθούν οι κρατούμενοι που στην ουσία είναι πολιτικοί κρατούμενοι των δημοσιογράφων και των ακτιβιστών. Και σύμφωνα με το θεμελιώδη δικαιώματα και το ε, πρωτογενές δίκαιο και τη στιγμή που το Αζερμπαϊτζάν έχει προσυπογράψει την Συμφωνία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και επειδή το Αζερμπαϊτζάν ανέλαβε ε, έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την περίοδο 2012-2013 θα πρέπει να αντιδράσει ανάλογα και να τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στα πλαίσια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και τώρα προχωράμε στους ομιλητές εξ ονόματος πολιτικών ομάδων, ο κύριος Πόσελτ από το ΕΛΚ. Κύριε Πρόεδρε, η ομάδα μας ε, είναι κατά τελευταίων όσων εδώ πέρα συνυπογράφονται. Κοιτάζουμε όλοι μαζί προς το Μπακού. Όχι επειδή ο κ. Σκέλεν είχε τραγουδήσει ο ίδιος πριν από 30 χρόνια στη Eurovision, αλλά επειδή το Αζερβαϊτζάν είναι σημαντικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέλος Συμβουλίου της Ευρώπης, της ΕΣΔΑ και άρα έχει περισσότερη υποχρέωση από άλλα κράτη-μέλη να τηρήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και το έκανε το Αζερβαϊτζάν εθελοντικά και το χαιρετίσουμε. Γι' αυτό θα αποδεχτεί, θα πρέπει να αποδεχτεί πώς θα κοιτάμε το τι θα κάνει. Και να σας πω κάτι το οποίο συνέβη πριν τον διαγωνισμό. Η κατεδάψη σπιτιών, η εκδίωξη ανθρώπων, η μη αποζημίωση, η έλλειψη κράτους δικαίου, ο ξυλοδαρμός διαδηλωτών, η καταπίεση της ελευθερίας του τύπου, της ελευθερίας ε, της θρησκείας. Αυτά δεν είναι αποδεκτά ακριβώς γιατί το Αζερβαϊτζάν για μας είναι σημαντικός εταίρος. Σας ευχαριστώ. Τώρα ο κύριος Ρέπο για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο διαγωνισμός της Eurovision ε, έχει τραβήξει την προσοχή των ΜΜΕ στο Αζερβαϊτζάν και οι άνθρωποι εκεί πέρα εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για να διαδηλώσουν στους δρόμους κατά της κατάστασής τους που είναι άθλια. Πολλοί άνθρωποι είναι στην φυλακή επειδή άσκησαν κριτική στην ε, κυβέρνησή τους. Η σκιά της απολυταρχίας ακόμη σκιάζει την ε, χώρα. Δεν υπάρχει μια δημοκρατική ε, να υπάρχει δημοκρατικό καθεστώς. Μπορεί λοιπόν το Αζερβαϊτζάν να αποτελέσει μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ όταν παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα των ίδιων των πολιτών του. Οι αρχές της χώρας αυτής ε, πρέπει να ανακαλέσουν τις διατάξεις περί δυσφήμισης από τον ποινικό κώδικα, να κάνουν εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις για την ελευθερία έκφρασης. Η υπηρεσία εξωτερικής δράσης πρέπει να απαιτήσει το Αζερβαϊτζάν να ερευνήσει όλες τις περιπτώσεις ε, περιορισμού της ελευθερίας έκφρασης και επίσης πρέπει να απελευθερωθούν οι πολιτικοί κρατούμενοι. Για τους φιλελεύθερους και δημοκράτες, ο κύριος Γιάννη Χερμπράντη για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στον Πακού τον προηγούμενο μήνα Ρώτησα τον πρόεδρο Αλίεφ για το ποια είναι τα σχέδιά του για να βελτιωθεί η κατάσταση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και των ΜΜΕ, της ελευθερίας δράσης των ΜΜΕ εν ώψη του, της Eurovision αυτή τη βδομάδα και μου απάντησε ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος για να βελτιωθεί η κατάσταση, διότι δεν είναι παρατέλεια δεν με εκπλήσει η, στάση του, διότι ο κόσμος ενδιαφέρεται στο Αζερβαϊτζάν λόγω του φυσικού αερίου, του, του πετρελαίου και των αγωγών φυσικού αερίου στο Ουσμπεκιστάν και στο Καζακστάν. Δεν μας ε, ενδιαφέρει ο λαός του Αζερβαϊτζάν και αν ο Επίτροπος Φούλε κατακρίνει την κατάσταση, ο πρόεδρος Μπαρόζο δύο εβδομάδες μετά δεν μίλησε ούτε μία φορά για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μιλούσε μόνο για θέματα ενέργειας. Άρα ποιο είναι το μήνυμά μας. Μη σας ενδιαφέρουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μας ενδιαφέρουν οι πηγές ενέργειας και τίποτα άλλο. Εάν λοιπόν είμαστε όμοιροι αυτής της κατάστασης, τότε δεν θα επέλθει καμία βελτίωση και μακροχρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προωθούσε καλύτερα και τα ενεργειακά της συμφέροντα αν ζητούσε μία ε, δημοκρατική πραγματικά κατάσταση παρά αν υποστηρίζει τον πρόεδρο Αλίεφ. Ε, εξ ε, της ε, Δημοκρατίας και την Ελευθερία για τις Ελευθερίες στην Ευρώπη, ο κύριος Πάσκα. Κύριε Πρόεδρε, το Αζερβαϊτζάν είναι μία χώρα η οποία συμμετέχει δραστήρια στην ε, Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και γίνονται και διαπραγματεύσεις σε σχέση με τη Συμφωνία Σύνδεσης Αζερβαϊτζάν Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένας πολύ σημαντικός οικονομικός μας εταίρος Γι' αυτό μας ενδιαφέρει και η πολιτική κατάσταση στη χώρα. Όταν όμως επιδεινώνεται η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι χρέος μας να ε, τονίσουμε στους εταίρους μας φιλικά ότι δεν μπορεί να γίνεται εκφοβισμός των ΜΚΟ, των δημοσιογράφων και ούτω καθεξής. Δεν είναι πολιτισμένα μέσα δράσης. Θα πρέπει λοιπόν να ε, υπάρχει ένα ε, σύστημα διπλωματικής προειδοποίησης έτσι ώστε το Αζερβαϊτζάν να δράσει σύμφωνα με τις διεθνείς επιταγές για τις δημόσιες ελευθερίες. Η ΕΕΔ θα πρέπει να βρει έναν τρόπο για να δει πώς θα μεταφέρει αυτό το μήνυμα. Και τώρα οι υπόλοιποι ομιλητές, καταρχήν η κυρία Κορχόλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, το Αζερβαϊτζάν είναι στο επίκεντρο των ΜΜΕ λόγω της Eurovision. Όμως η προσοχή αυτή είναι αρνητική λόγω των προβλημάτων στα ανθρώπινα δικαιώματα. Περιορίζεται η δουλειά των ΜΚΟ, δημοσιογράφοι, χρήστες κοινωνικών μέσων έχουν ε, φυλακιστεί. Η κυβέρνηση έχει πει πολλά, έχει δώσει πολλές προσχέσεις για βελτίωση της ε, κατάστασης, ε, για αλλαγή της νομοθεσίας. Υπάρχει μια νέα επιτροπή που εξετάζει τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά αυτή η επιτροπή πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Το Αζερβαϊτζάν είναι μια χώρα στην πολιτική γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και πρέπει βεβαίως να δρά καλή την πίστη. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο έχει η κυρία Κρέτσου. Ευχαριστώ. Πολύ χρήσιμη αυτή η πρόταση ψηφίσματος, διότι προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Αζερβαϊτζάν και ελπίζω ε, οι Αζέροι να, τηρήσουν, να τηρήσουν τις ε, διεθνείς συμφωνίες τις οποίες έχουν ε, προσυπογράψει. Ένα τέτοιο πολιτιστικό γεγονός έχει συμβολικό χαρακτήρα και δεν πρέπει να ξεχνάμε την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μας απασχολεί και μας ανησυχεί η κατάσταση δίωξης των δημοσιογράφων και το γεγονός ότι απαλωτριώθηκαν μεγάλες εκτάσεις και εκδιώχθηκαν οι άνθρωποι από τα σπίτια τους. Δεν έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης και συνέρχεστε και τους συνέρχεστε, γι' αυτό θα πρέπει να τηρηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να προωθεί το ζήτημα αυτό η ΕΕΔ. Έχετε μια μπλε κάρτα Κυρία Κρέτσου, δέχεστε το ερώτημα. Ωραία. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κυρία Κρέτσου, θα ήθελα ε, να σας ρωτήσω το εξής. Φυσικά είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά τα ζητήματα που εγείρετε, αλλά ήθελα να ρωτήσω αν πιστεύετε πως είναι δικαιολογημένο αυτό το κατεπήγον ζήτημα, δεδομένου του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και το Αζερβαϊτζάν συμμετέχουμε σε διάφορες διεθνείς πλατφόρμες και οργανισμούς όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης. Το ζήτημα αυτό έχει συζητηθεί επανειλημμένα. Πιστεύετε ότι με αυτό το ψήφισμα θα λύσουμε το πρόβλημα? Όταν μιλάμε για το ότι πρέπει να σώσουμε ζωές, Νομίζω ότι ποτέ δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ νωρίς ή πολύ αργά. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή τη χώρα και να την εντάξουμε στο ευρωπαϊκό σύστημα αξιών και τίποτα δεν δικαιολογεί τα τεκτενόμενα στο Αζερβαϊτζάν την παρούσα στιγμή. The next speaker is Η κυρία για λεπτό. Ευχαριστώ με την ευκαιρία αυτή με το θέμα ε, του επίγοντος να μιλήσω για το, για το στάτους αυτών των ε, προτάσεων επίγοντος. Όταν μιλήσαμε για εμπορικές συμφωνίες και όταν λέγαμε ότι θα πρέπει το Αζερβαϊτζάν να είναι μη είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, ήμασταν σοβαροί. Πόσο σοβαροί είμαστε όταν μιλάμε για ενεργειακά προγράμματα τα οποία είναι ισόφελός μας. Δηλαδή έτσι είμαστε αποδοτικοί τη στιγμή που δεν συμβαίνει τίποτα ως προς την προάσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μιλάμε για θέματα στα οποία δεν δόθηκε λύση, αποτέλεσαν αντικείμενο άλλων ψηφισμάτων και νομίζω ότι το Αζερβαϊτζάν δεν τηρεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες προδιαγραφές και μία συνοχή ως προς τον τρόπο που θίγουμε ορισμένα ζητήματα για να είμαστε αξιόπιστοι. Μην μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά να μιλάμε για, ενεργειακές, για συμφωνίες στον ενεργειακό τομέα εις όφελος του Ευρωπαίου πολίτη. Χρήσιμη αυτή η συζήτηση, αλλά θα πρέπει να γενικευθεί και να δούμε ποια είναι τα κριτήριά μας σε σχέση με τις ε, συμφωνίες σύνδεσης. Κυρία Νίκολαη, ο κύριος Πόσελτ ε, θα ήθελε να σα υποβάλει ένα ερώτημα. Μπλε κάρτα, δέχεστε, ναι. Κυρία Νικολάη, γνωρίζετε πως δεν είμαστε διπλωμάτες ούτε επιχειρηματίε. Είμαστε βουλευτές με πρώτο καθήκον τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και Συνεργαζόμαστε με πολλές χώρες, με τη Ρωσία, με την Ουκρανία, με πολλές χώρες εταίρους. Και πάντα πρέπει και τους υπενθυμίζουμε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Uh, Συμφωνώ κύριε Πόσελτ, αλλά ναι. εσείς ψηφίσατε υπέρ της Συμφωνίας Σύνδεσης με το Αζερμπαϊτζάν γιατί είχαμε θέσει ως πρόκριμα την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν θα πρέπει να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. the Ευχαριστώ. Περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Εφτά συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο. Περνάμε στην κυρία Εσαγιά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι ικανοποιημένη με το γεγονός πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει την άποψή του για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερβαϊτζάν. Έχουν μια πολύ καλή ε, διαφημιστική εκστρατεία στο πλαίσιο του διαγωνισμού της Eurovision αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουν γίνει πολλά πράγματα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η διεθνής κοινότητα κάνει τα στραβά μάτια. Τώρα ασκούμε κριτική στη χώρα, αλλά η κριτική δεν επιτρέπεται εντός της ίδιας της χώρας. Λογοκρισία, και υποφέρουν ε, οι πάντες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Γιακονσάρη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την Σάρη Εσαγιά, καθώς και άλλες, ε, άλλους συναδέλφους. Ε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ψήφισμα είναι σημαντικό δηλαδή το Κοινοβούλιο να καλέσει τις οικίες αρχές να απελευθερώσουν τους πολιτικούς κρατουμένους. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να παρακολουθήσει τις εξελίξεις κυρίως μετά τον διαγωνισμό Eurovision ο διαγωνισμός τραγουδιού Eurovision είναι μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν στη διοργάνωση της Eurovision. Και ξαναλέω ότι είναι σημαντικό να μην ζουν όλοι μέσα στο φόβο. Σας ευχαριστούμε κύριε Σφουτσόφσκι. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Υποστηρίζω την πρόταση ψηφίσματος. Μας ενδιαφέρει η μοίρα του Αζερμπαϊτζάν γιατί είναι καταπληκτική η ιστορία και οι παραδόσεις ε, της χώρας αυτής. Ε, προσπαθεί δεν να προσχωρήσει στην ευρωπαϊκή οικογένεια, συμμετέχει σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, τώρα διοργανώνει τον ε, διαγωνισμό Eurovision. Αλλά αν θέλει να ακολουθήσει την ίδια ρότα με την Ευρώπη, οφείλει να συμμορφωθεί και με τα πρότυπα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εδώ δεν έχει καλές επιδόσεις. Ε, ήρθε η στιγμή λοιπόν να θίξουμε αυτό το ζήτημα και να απευθύνουμε έκκληση προς τις αζερικές αρχές, ε, κυρίως όταν τα φώτα της δημοσιότητας θα πέσουν πάνω σε αυτή τη χώρα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ο κύριος Βατσικόφσκι. Νομίζω πως το συμπέρασμα είναι απλούστατο. Τα τελευταία 20 χρόνια από την ανεξαρτησία και μετά βλέπουμε πως η οικονομική πρόοδος έχει επιτευχθεί. Είναι μια οικονομική τίγρης η χώρα, αλλά βεβαίως η πολιτική πρόοδος δεν ακολουθεί την οικονομική. Λείπουν πολλά ακόμα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικά όταν μιλάμε για ελευθερία του λόγου. Έχουμε πολλά παραδείγματα περιφρόνησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πάντα πρέπει να υψώνουμε τη φωνή μας υπέρ ε, των δημοσιογράφων που δεν μπορούν να μιλήσουν ελεύθερα, που κατηγορούνται και φυλακίζονται Υπήρξε παράδειγμα δημοσιογράφου, ο οποίος μετά από δύο άρθρα σε τοπική εφημερίδα καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκιση. Πράγματα απαράδεκτα. Είναι ατυχές ε, το ότι δεν μιλήσαμε στον Πακού στη διάρκεια της Συνόδου. Ο επόμενος συμβολητής είναι ο κύριος Κυρίλοφ. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία έχουν μεγάλη σημασία στη γειτονιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν υπάρχουν κατεπήγοντες λόγοι, δεν θα πρέπει ε, να μας απασχολούν τα πράγματα αυτά στα κατεπήγοντα. Ναι, το είπαν στην άλλη. Πράγματι υπάρχουν στην περίπτωση του Αζερβαϊτζάν κάποια προβλήματα, αλλά ποιο είναι το κατεπήγον, η Eurovision. Ε, οι συνάδελφοι λένε πως ε, οι αρχές ίσως καταστήλουν τους αντιπάλους τους μετά της ε, μετά το διαγωνισμό. Μα αυτό το ψήφισμα θα το δεχτούν ως ε, πισόπλατο μαχαίρωμα οι αρχές ε, του Αζερβαϊτζάν. Θα γίνει μια συζήτηση στην Ολομέλεια με τον Επίτροπο, τον κύριο Φίλε. Έτσι θα έχουμε αποτελέσματα, καθώς είμαι σίγουρος πως οι αζερικές αρχές θα γνωρίζουν το κείμενο του ψηφίσματος αυτού. Σας ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής. Α, μια μπλε κάρτα. Από τον κύριο Πόσελτ. Question, yes. You have the floor. Δέξτε το ερώτημα, ναι. Κύριε Κυρίλοφ, γνωρίζετε πως ολόκληρη αυτή τη βδομάδα πριν από τη Eurovision βγήκαν διαδηλωτές και ξυλοκοπήθηκαν αγρίως στους δρόμους Και οι άνθρωποι αυτοί βεβαίω ε, θα εκπλήσονταν ε, αν μάθαιναν πώ δεν το θεωρείται αυτό κατεπήγον και περιμένετε να μπουν φυλακοί. Ναι, ναι. Τα παρακολουθώ τα γεγονότα στη χώρα. Αυτό το οποίο είναι ενδιαφέρον διάβασα σήμερα στην International Herald TV πως χτες έγινε ειρηνική διαδήλωση κατά του καθεστώτος ε, χωρίς άδεια και πέρασα από τους κεντρικούς δρόμους. Πρέπει να τα συζητήσουμε ορισμένα πράγματα σοβαρά με τις αρχές. Ε, αλλά αυτό το οποίο λέω εγώ κύριε Πόσελτ είναι πως δεν είναι αυτός ο τρόπος. Μα κοιτάξτε πώς είναι μέσα στην αίθουσα. Δεν είναι τρόπος αυτός για να ασχοληθούμε με μια χώρα η οποία είναι πολύ σημαντική σε στρατηγική ε, γειτονιά της Ένωσης. Σας ευχαριστώ κύριο Σκούκαν. Σας ευχαριστώ η προστασία και η περάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η προστασία του κράτους δικαίου, του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθε, το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης συνιστούν βασικά ε, θεμελιώδη δικαιώματα και το ίδιο ισχύει και για τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για το Αζερβαϊτζάν. Προτείνω να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις και αν χρειαστεί μπορούμε τότε να απευθύνουμε επικρίσεις κατά της χώρας. Δεν νομίζω καν να ενδιαφερθεί κανείς το Αζερβαϊτζάν ούτως ή άλλως για τις επικρίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θα έπρεπε επίσης να συζητήσουμε ζητήματα όπως η καταστολή των ειρηνικών διαδηλώσεων, φυλάκιση δημοσιογράφων ή ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να ρυθμιστούν το ταχύτερο δυνατόν και είναι το ελάχιστο που μπορούμε να ζητήσουμε από το Αζερβαϊτζάν που φιλοδόξει να έχει αυτή την εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα πρέπει να εγκρίνουμε το ψήφισμα. Ευχαριστώ η κυρία Άννα Γκόμε Ο πρόεδρος Μπαρός, πήγε στον Μπακού, αλλά δεν μίλησε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε για την επιδείνωση της κατάστασης, παρά, όλες, παρά όλα τα υπεσχημένα περί μεταρρυθμίσεων κτλ. Υπάρχουν απειλές καταστολή ειρηνικών διαδηλώσεων, φυλάξει δημοσιογράφων ε, και όλα αυτά συμβαίνουν κάτω από το φω τη δημοσιότητας ε, του διαγωνισμού Eurovision. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιδιώξει συγκεκριμένου στόχους, δημοκρατικές μεταρρυθμίσει, εφαρμογή της συμφωνίας ω προς την ελευθερία έκφραση. Ε, και άλλες θεμελιώδεις ελευθερίες. Ε, επίσης θα έπρεπε να συνοδεύεται αυτή η δράση με επιβολή κυρώσεων από πλευράς μας. Ευχαριστούμε και ας ακούσουμε τώρα τον Επίτροπο Ποτόσνικ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Αζερμπαϊτζάν έχουν σχέσεις που όμως δεν έχουν εξαντλήσει ε, το δυναμικό τους. Η Οικονομική ε, Ένωση των δύο εταιρών ε, θα καταστεί δυνατή μόνο αν το Αζερβαϊτζάν ε, κάνει μεγαλύτερες προσπάθειες ως προς τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις εκλογικής διαδικασίας, προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος και συναφή ζητήματα. αυτό αποτυπώνεται στο ψήφισμα της 15ης Μαΐου Μαΐου του Κοινοβουλίου. Το Μάρτιο υπήρξαν ειρηνικέ διαδηλώσει και ακολούθησε καταστολή, κυρίω όταν μιλάμε για τη διαδήλωση των Πακού στι 2 Απριλίου. Αυτό ε, συνιστά σοβαρό κόλλημα ε, στην όλη διαδικασία δημοκρατική μεταρρύθμισης και δεν συνάδει με τα υπεσχημένα από πλευρά του Αζερβαϊτζάν ε, στα πλαίσια των δεσμεύσεων της χώρας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα πλαίσια του ΑΣΑ. Ο Μιτσίτλη απελευθερώθηκε ήδη και ελπίζω στις 28 Μαΐου να απελευθερωθούν και άλλοι πολιτικοί κρατούμενοι συχνά. Ε, παραβιάζονται τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα με υποχρεωτικές εξώσεις ε, παρά, ε, το αντίθετε, παρά την ύπαρξη αντίθετων δικαστικών αποφάσεων και χωρίς καμία προειδοποίηση. Στις 27 Φεβρουαρίου υιοθετήθηκε νέο νομοσχέδιο ή μάλλον νέο υπουργικό διάταγμα αλλά αναρωτιόμαστε αν η νέα νομοθεσία θα βελτιώσει την κατάσταση. Αναφέρθηκαν πολλοί στο διαγωνισμό τραγουδιού ε, Eurovision. Να, λοιπόν, ένα παράθυρο ευκαιρίας για τις οικίες αρχές όμως φαίνεται ότι δεν άδρεξαν την ευκαιρία. Στις 16 Μαΐου η διάσκεψη για την ελευθερία των ΜΜΕ που διοργανώθηκε από ε, την εκστρατεία τραγουδίστρια για τη δημοκρατία Sing for Democracy ε, ανέφερε ότι σε μεμονωμένες περιπτώσεις καταγγελιών διεξάγεται ακόμη η έρευνα όπως στην περίπτωση Καντία Ισμαήλοβα που ήταν μια ερευνητική δημοσιογράφος ε, που ε, υπέστη εκβιασμό. Επίση, στι 16 Μαΐου υπήρξαν δράσεις της αντιπολίτευσης και ακτιβιστέ συνελήφθησαν αλλά απελευθερώθηκαν στη συνέχεια 16 χιλιόμετρα έξω από τον Πακού. Ε, το περιβάλλον για τα ΜΜΕ χαρακτηρίζεται από αυτό λογοκρισία και περιορισμό των δημοσιογράφων. Πρόσφατα παραδείγματα είναι κράτηση δύο δημοσιογράφων σε μια περιφερειακή πόλη του Αζερβαϊτζάν. Το ίδιο συνέβη για δημοσιογράφους που κατηγορήθηκαν ότι κατασκόπευαν από πλευράς του Ιράν. Ε, και ε, η επίσκεψη του Επιτρόπου Φίλε στην Αζερμπαϊτζάν στα πλαίσια της σύσκεψης Euronest έδωσε τη δυνατότητα να εκφράσουμε τις αυξανόμενε ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τονίζουμε την ανάγκη να, ε, τηρήσει τις δεσμεύσεις του το Αζερμπαϊτζαν στα πλαίσια της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Αζερμπαϊτζάν, όπως ξέρετε, έχουν μια πολύ ολοκληρωμένη και πλούσια η αδημερή ατζέντα, η βασική αρχή από τις οποίες εδράζεται οποιαδήποτε σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτη χώρα είναι ο σεβασμός ε, του κράτους δικαίου της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, αν αυτό διακυβευτεί τότε η περιφερειακή μας συνεργασία στερείται πλέον νοήματος. Επικρατεί μεγάλη διαφάνεια σε σχέση με την αξιολόγηση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε οποιαδήποτε χώρα και όπως σας είπα η έκθεση πρόοδου που εξεδόθη το Μάιο αποτυπώνει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αυτής. Τέλος, η πλήρης εφαρμογή της ευρωπαϊκής, του σχεδίου δράσης για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας αναμένεται. Η πολιτική κρατούμενη όντω θα πρέπει ε, να απελευθερωθούν και η ελευθερία έκφρασης και ε, συγκέντρωσης θα πρέπει να κατοχυρωθούν. Ο ειδικό εισηγητής της του Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου τη Ευρώπη για του πολιτικού κρατουμένου, ε, ούτω ή άλλω παρακολουθεί τι εξελίξει και μα ενημερώνει. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Έχουμε λάβει έξι σχέδια ψηφίσματο για να κλείσει αυτή η συζήτηση. Πέρα λοιπόν και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί μετά το πέρας όλων των ε, κατεπηγόντων συζητήσεων της απογευματινής συνόδου. Περνούμε τώρα στην